εγκρίνονται αυτοί οι διορισμοί. Η διάσκεψη των Προέδρων, κυρίε και κύριοι, έχει τι εξή προτάσει ε, για την διεξαγωγή των εργασιών μα ε, για το 2013. 14η μέχρι 17η Ιανουαρίου, 4η έω 7η Φεβρουαρίου, 11η έω 14η Μαρτίου, 15η έω 18η Απριλίου, 20η έω 23η Μαΐου, 10η έω 13η Ιουνίου, 1η έως 4η Ιουλίου, 9η έως 12η Σεπτεμβρίου, 7η έως 10η Οκτωβρίου, 21η έως 24η Οκτωβρίου, 18η έως 21η Νοεμβρίου, 9η έως 12η Δεκεμβρίου αυτές οι περίοδοι συνόδου. Οι προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογιών σε αυτές τις προτάσεις ε, είναι η 3η 15η Ιανουαρίου 19.00 ώρα. Η ψήφιση θα γίνει την Τετάρτη. Περνάμε σε μια νέα διαδικασία. Έχουμε τρεις προτάσεις ε, από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 70α του κανονισμού για την ε, έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων και την εντολή για τρεις νομοθετικές διαβουλεύσεις. Η σειρά αυτών των οι, τα αιτήματα έχουν ε, μεταφραστεί στις γλώσσες και μπορούν να ε, αντληθούν από